θα σημάνει πολλά όχι μόνο για τη ζωή των ανθρώπων που βοηθούμε αλλά και για το στάτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 12, έληξε συζήτηση. Πάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Σάρμπου αναγνώριση της Γεωργίας ως στρατηγικό τομέα για την επισητιστική ασφάλεια. Για τέσσερα λεπτά η συγγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω την έκθεση αυτή που αναφέρεται στη Γεωργία γιατί ο Γεωργίας τελικά ε, η Γεωργία τελικά ε, έχει αγνοηθεί επανειλημμένα ως στρατηγικός τομέας της Ένωσης. Ή, αυτό είναι λάθος. υπάρχουν καινούριε προκλήσεις. Υπάρχει η κλιματική αλλαγή που μειώνει συνεχώς τα επιστημιστικά αποθέματα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τουλάχιστον 70% πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων τα επόμενα μέχρι το 2050 για να μπορέσει να εξασφαλιστεί πλήρης ε, επιστημιστική ασφάλεια για όλους. Ε, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει κάποια ε, να φροντίσει κάτι να κάνει. Πρέπει να έχουμε μια γεωργία που θα εξασφαλίζει την, ε, θα παρέχει επιστημιστική ασφάλεια και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αλλά και για τον κόσμο βέβαια ολόκληρο. Δεν μπορούμε να μιλούμε για επισκεπτική ασφάλεια βεβαίως αν δεν επιλύσουμε δύο βασικά προβλήματα. Τη πτυτικότητα των αγορών και των τιμών και εδώ θα ήθελα να πω ότι ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα πλαίσια της καινούργιας κοινή αγροτικής πολιτικής να ενοποιηθεί ο ρόλος των εργαλείων που υπάρχουν για την ρύθμιση των αγορών και των τιμών. Αυτή τη στιγμή η, τα αποθέματα τροφίμων είναι πολύ μικρότερα από ό,τι ήταν παλιά και από ό,τι λέγεται καλύπτουν τις ανάγκες ε, του κόσμου μόνο για 1,5 μήνα. Θα πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να δημιουργεί αποθέματα αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να ε, δούμε πρώτα πρώτα τις τιμές. Εμάς περιπτώσει τα αποθέματα αυτά θα πρέπει να είναι διεθνή, να ε, ρυθμίζονται σε διεθνέ επίπεδο αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει την πρωτοβουλία για το θέμα αυτό και ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε και και στην έκθεση είναι η κατάσταση των νέων γεωργών αν μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τους νέους γεωργού μόνο 7% των γεωργών είναι κάτω από 30 ετών αυτή τη στιγμή στη, στη γεωργία, στο γεωργικό τομέα. Εμείς αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή γεωργία θα πρέπει να προσελκύσουμε περισσότερα νέα άτομα στον τομέα αυτό, να βοηθήσουμε στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων εκμεταλλεύσεων, μικρών εκμεταλλεύσεων, βιολογική γεωργία κτλ. Να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν, που μπορούν να στηρίξουν την εναλλακτική γεωργία και για... δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχει φτώχεια και πείνα και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το χειμώνα που μας πέρασε ε, πολλές χιλιάδες Ευρωπαίων βοηθήθηκαν από τη ε, επισητιστική βοήθεια που δόθηκε. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης συγητές και όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας για την καλή δουλειά που έκανα και τη συνεισφορά τους. Να ευχαριστήσω επίσης και τη γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας και ελπίζω πραγματικά αύριο να κάνουμε την να υπερψηφιστεί έκθεση αυτή που θα βοηθήσει τους πολίτες μας. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρμπό για την εξαιρετική τη εργασία για την έκθεση αυτή, καθώς και για τη συνεργασία της με όλους τους κοιόδης. Ακολουθεί μια εργασία που είχα αναλάβει στην προηγούμενη θητεία. Και λυπάμαι γιατί μόλις λίγο πριν τα μεσάνυχτα συζητάμε το θέμα αυτό και ίσως πράγματι να βρισκόμαστε στο παραπέντε με την κατάσταση αυτή. Η έκθεση λοιπόν είναι πολύ χρήσιμη και στα πλαίσια ιδιαίτερα της συζήτησής μας για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Τις ανησυχίες που είχα να εκφράσω τις λέει και το ίδιο το κείμενο. Η ίδια η ιδέα ότι ένα σύστημα είναι καλύτερο από άλλο είτε πρόκειται για οργανικό, βιολογικό είτε για το εντατικό είναι λανθασμένη. Πρέπει να τα δούμε όλα μαζί και δεν νομίζω ότι έχουμε όλες τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Το κύριο πρόβλημα με τη γεωργία είναι τα χαμηλά εισοδήματα των γεωργών. Οι νέοι ιδίω γεωργοί δεν δέχονται να εργαστούν δωρεάν και πρέπει να το θέσουμε αυτό το θέμα κάποτε. Ευχαριστώ για την έκθεση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι συνεχής η αύξηση του πληθυσμού και γι' αυτό χρειάζεται όλο και εντατικότερη εκμετάλλευση της γεωργίας για την παραγωγή ταροφίμων. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε και μεγαλύτερη διαφάνεια στην παραγωγή της τροφιμικής αλυσίδας και διασφάλιση των εσόδων των αγροτών και αγροτισών. Προσωπικά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμοστεί μια στεναρή πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου που να καταλήξει στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτής και την συνέχιση της δραστηριότητας των γεωργών. Η γεωργία έχει ιδιαίτερη σημασία ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες και καθυστερημένες περιοχές και πρέπει να τους χορηγήσουμε κίνητρα για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους οι γεωργοί καθώς και να προσελκυστούν περισσότεροι κάτοικοι στην Ήπεθρο ο κύριος Λουίς Άλντες. Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ ειλικρινά την κυρία Σάρμπου για την εξαιρετική της έκθεση και το ελπίζω το Συμβούλιο να τη λάβει υπόψη της Να λάβει υπόψη λοιπόν το Συμβούλιο και η Κομισιόν αυτή την έκθεση ούτως ώστε να μην τέθει το ζήτημα μόνο από γεωργικής πλευράς αλλά να εξεταστεί και οικονομική, δημοσιονομική και ανθρωπιστική του πτυχή. Οι φιλόδοξοι στόχοι της ΚΑΠΑ θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνο αν η μεταρρύθμιση αυτή ξεπεράσει τα όρια της Γεωργίας. Αν δηλαδή οριζόντια ληφθούν οι υπόψεις στις άλλες, και στις άλλες πολιτικές συνολικά. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Też przyłączam się do gratulacji dla pani Sarbu za znakomite sprawozdanie ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που συνεχάρισαν την κυρία Σάρμπου για την έκθεση αυτή. Είναι πολύ σημαντική. Ε, ίσως από τις πιο σημαντικές της θητείας μας. Ο πληθυσμός της γης γίνεται όλο και μεγαλύτερος και τα τρόφιμα είναι ε, ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η... Γιατί η τροφή ε, είναι κάτι που δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές μορφές τροφής. Και μέχρι τώρα βρούσαμε με, σαν να βρισκόμαστε σε ε, περίοδο παχαίων αγελάδων και, και πλεονασμάτων στον επισητιστικό τομέα. Τώρα βλέπουμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, να προστατεύσουμε την ε, παραγωγή, τη γεωργία για να έχουμε επιστηστική ασφάλεια. Κύριε Πρόεδρε, όπως συμβαίνει και στη, σε άλλους τομείς και στην πολιτική δεν ε, συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι κάτι όταν το έχουμε μόνο αν δεν το έχουμε αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε τη σημασία του θα πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη να σκεφτούμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κάτι τέτοιο με, την, με τα τρόφιμα και Πράγματι πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας για να αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε, να υπάρχει επιστηστική ασφάλεια για όλους. Θα πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική της, στη Γεωργία για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στους πολίτες της Ευρώπης ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή, η άνοδος των τιμών, όλα αυτά επηρεάζουν το, την επιστηστική ασφάλεια της Ευρώπης και γι' αυτό πρέπει να δράσουμε τώρα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Σταμπάτσι. η επισητιστική ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών θα αποτελέσει και το τη μεγαλύτερη πρόκληση στα επόμενα χρόνια διότι τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό θα γίνουν εξίσου πολύτιμα όπως και το πετρέλαιο σήμερα. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη αυτή η έκθεση διότι ξεκινάμε την προετοιμασία των συζητήσεων για το μέλλον της ΚΑΠ και τις πρώτες συζητήσεις για τις δημοσιονομικές προπτικές. Και μερικοί θα ήθελαν να αρχίσουν να περικόπτουν τις ε, γεωργικές δαπάνες η γεωργία όμως δεν μας παρέχει μόνο τρόφιμα αλλά και αξίες που είναι αναντικατάστατες. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η επισητιστική ασφάλεια για μένα είναι ένα... Ε, ε, ε, μου δημιουργεί πρόβλημα στην έκθεση όταν θεωρείται ότι όλα τα κράτη την αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο τρόπο. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω δύο πράγματα. Πώς είναι δυνατόν σε μία χώρα με πολύ καλές συνθήκες για τη γεωργία έχουμε παιδιά και ενήλικες οι οποίοι πεινάνε. Πώς είναι δυνατόν η γεωργία αναπτυσσόμενη με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται με την εντατική γεωργία και που παρέχει ε, ε, για την παροχή πρώτης ύλη στη βιομηχανία. Γιατί λοιπόν αυτά τα γεωργικά προϊόντα μεταποιούνται στο εξωτερικό και επανισάγεται μετά το τελικό προϊόν στη χώρα μας με υπερβολικές τιμές. Ο κύριος Κέλλη. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Σάμπου για την εξε... εξαιρετική δουλειά που έκανε. Κάλυψε πολλές πτυχές, αλλά θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη για μια καινούρια κοινή αγροτική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσει να μην απαξιωθεί η ΚΑΠ. Επίσης θα πρέπει να βοηθηθούν οι νέοι γεωργοί να, που θα μπουν στον τομέα. Ε, ίσως αυτή τη στιγμή μάλλον έχουμε μια πολιτική η οποία ευνοεί την καλλιέργεια ενεργειακών προϊόντων όταν αρχίζουν και λείπουν τρόφιμα. Μήπως πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την πολιτική μας πριν τα πράγματα θα σου σε άσχημο σημείο. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη, ο κύριος Σαντζέντη. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την έκθεση ανακαλύπτουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στη Γεωργία όπως σήμερα. Δεν μπορούμε εμείς ε, να μεταφέρουμε προϊόντα από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Δεν θα μπορούμε πια να εισάγουμε μήλα και πάπρικα από τη Βραζιλία και από την Κίνα. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε κρέατα διότι όλα αυτά τα προϊόντα ταξιδεύουν για βδομάδες και χρησιμοποιούνται συντηρητικά και κόντρα συντηρητικά τα οποία είναι ιδιαίτερα νοσηρά για τον άνθρωπο. Μετά εμείς εκπλησόμαστε να βλέπουμε αρρώστιες, όγκους, καρκίνους που εμφανίζονται. Πρέπει λοιπόν εμείς να υποστηρίξουμε τις μικρές εκμεταλλεύσεις και οι οποίες μας βοηθούν να βγαίνουμε από την κρίση στην Ευρώπη. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικός τομέας στον επισητισμό δεν θα μπορέσουμε, δεν θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την επισητιστική κυριαρχία. Όσο μια χώρα είναι περισσότερο ανεξάρτητη στον επισητιστικό τομέα, τόσο πιο δύσκολα μπορεί να ταΐσει τους πολίτες του. Η επισητιστική λοιπόν κυριαρχία έρχεται να καταπολεμήσει αυτή την έλλειψη τροφίμων η οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και αυτό κυρίω λόγω της ε, κερδοσκοπίας, της ε, χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας στον τομέα των τροφίμων. Για να αποφύγουμε λοιπόν την κερδοσκοπία πρέπει να σταματήσουμε με τα παράγωγα ε, και άλλα νοσηρά προϊόντα τα οποία οδηγούν στην κερδοσκοπία. Ο πώς το αναγνωρίζει δηλαδή και η έκθεση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα στην τροφή. Σήμερα συζη... που... συζητούμε ε, το θέμα της γεωργίας το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο σπάνια συζητιέται εδώ συζητάμε χίλια δυο άλλα θέματα συζητάμε τους στοχούς της Ευρώπης τους Ρωμά συζητάμε τα συζητήσαμε αυτά στις αρχές της ε, Ουγγρικής Προεδρίας αλλά για τους ανθρώπους αυτούς το φαΐ στο τραπέζι είναι το, βασική, το βασικό τους μέλημα σε αυτή τη ζωή. Η, όπως το είπαν και άλλοι, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα, τα τρόφιμα και την επιστημική ασφάλεια για τις μελλοντικέ γενιές αν θέλουμε να φτιάξουμε μια σωστή Ευρώπη. Κυρία Τζουτζέβα, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση αυτή, η οποία είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, γιατί αυξάνονται πάρα πολύ οι τιμές της στα τρόφιμα και επειδή ε, και λόγω φυσικών καταστροφών αλλά και λόγω της τιμής ενεργειακών προϊόντων και του, του πετρελαίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ασχολήθηκαν με την έκθεση αυτή. Η επιστημιστική ασφάλεια είναι απαραίτητη για το ένα, για τα εκατομμύρια εκείνων των ανθρώπων που ακόμη ε, πεινάνε για την Ευρώπη η κοινή αγροτική πολιτική ε, κάνει τη διαφορά όμως επικρίθηκε επανειλημμένα η πολιτική αυτή αλλά μέχρι τώρα κατάφερε να εξασφαλίσει να εγγυηθεί επισητιστική ασφάλεια στην Ευρώπη και μάλιστα σε λογικές τιμές η επισητιστική ασφάλεια είναι από τις λέξεις κλειδιά στην ανακοίνωση που κάναμε το που υιοθετήσαμε τον Νοέμβρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γεωργία με ορίζοντα το 2020. Η έκθεση αυτή που συζητούμε τώρα τονίζει ιδιαίτερα το θέμα της τεράστιας μεταβλητότητας των τιμών που σχετίζεται βεβαίως με την επιστημιστική ασφάλεια η Κομισιόν συμφωνεί απόλυτα ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταπολεμηθεί η, η μεταβλητότητα, ε, η αστάθεια των τιμών. Βεβαίως πρέπει να δούμε θέματα που σχετίζονται με την αγορά, αλλά αυτό και εδώ πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει διαφάνεια. Η έκθεση συνίσταται, ε, συστήνει συγγνώμη, τη δημιουργία ενός διεθνού τροφιμικού συστήματος με διεθνή αποθέματα δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει Γι' αυτό χρειάζεται να συζητηθεί περαιτέρω, να αναλυθούν περισσότερο οι εμπειρίες του παρελθόντος. Ε, το 2008 λόγου χάρη υιοθετήσαμε αυτό το μέσο το, το, το ενός δις σε σχέση με τα τρόφιμα. Ποια ήταν τα αποτελέσματά του. Θα πρέπει να τα δούμε λοιπόν αυτά για να... Ε, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε θα πρέπει να επέμβουμε και να φροντίσουμε και για τις τιμές και πραγματικά το G20 θα ασχοληθεί με το θέμα των τροφίμων και των αποθεμάτων τροφίμων και βεβαίως θα εμπλακεί έντονα τις επόμενες εβδομάδες σχετικές συζητήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος πολλοί από εσά ζήτησαν να υπάρχει μια ισχυρή αγροτική πολιτική και πολιτική της υπαίθρου εδώ στην Ευρώπη να, για να βοηθηθούν οι αγρότες για να μπορέσουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Η Κομισιόν συμφωνεί απόλυτα με αυτό Δεν υπάρχει καλύτερο εργαλείο στη διάθεσή μας από μια ισχυρή αγροτική πολιτική, πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και όπως είπαν και πολλοί από εσά, θα πρέπει να φροντίσουμε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στο γεωργικό τομέα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Η επόμενη Ολομέλεια, 18 Ιανουαρίου από τις 9 στη 1, από τις 3 στις 8.